κυβερνήσεων να ε, αρθούν στο ύψο των περιστάσεων, πράγμα που δεν του χαρακτηρίζει το τελευταίο διάστημα. Ευχαριστώ κύριε Πεγιό. Ε, ολοκληρώνεται η συζήτηση, η ψηφοφορία θα ακολουθήσει στι 12. Επόμενο θέμα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, είναι η έκθεση του κυρίου Κύριλοφ με θέμα την αναγκαιότητα μια στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Νότιο Κάφκασο. Ο εισηγητή έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πίτροπε Φούλε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και όλους τους εισηγητές και όσους συναδέλφους πήραν μέρος στην επεξεργασία αυτής της σημαντικής έκθεσης για τον Νότιο Κάυκασο δεν είναι μόνο μια κοντινή περιοχή, αλλά έχει και πολύ στρατηγική σημασία γενικότερα στον τομέα της ασφάλειας. Γι' αυτό ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να πάρει μέρος ενεργά στη σταθεροποίηση της περιοχής, να οδηγήσει χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία στη σταθερότητα και στις ειρηνικές σχέσεις υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες τις πρωτοβουλίες που αυξάνουν και τονώνουν την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή μέσω της ανατολικής εταιρικής σχέσης και περαιτέρω περιφερειακής συνεργασίας ειδικών ρυθμίσεων για, τη, για την ελεύθερη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ χωρίς θεωρήσεις είναι προς το ζωτικό σαφέρον και των τριών αυτών χωρών και των δικών μας χωρών να συνεχίσουν στην οδό του εκδικρατισμού. Το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κυρίαρχα χαρακτηριστικά για τον καθορισμό των μελλοντικών του σχέσεων με την Ένωση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να παρέχει λοιπόν τεχνική συνεργασία έτσι ώστε να προωθήσει γενικότερα τη δημοκρατία στην περιοχή αυτή. Ο ρόλος των χωρών αυτών σε επίπεδο περιοχής θα έλεγα συνδέουν την Κασπία και την Κεντρική Ασία με την Ευρώπη και γι' αυτό η στρατηγική σημασία τους αυξάνεται συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα που αφορούν την ενέργεια στην περιοχή, όπως το πρόγραμμα του δικτύου ε, του αγωγού Ναμπούκο. Τα προβλήματα που εκκρεμούν στη Γεωργία και στον Αγκόρνο Καραμπά είναι εμπόδια για τον πλήρη εκδημοκρατισμό και την κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη. Μόνο το 2008 με την πολεμική σύραξη στη Γεωργία μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνειδητοποιήσει τον σημαντικό ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει στην περιοχή. Ακριβώς λοιπόν η συνειδητοποίηση αυτή και η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας δίνει τις δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει με πιο ενεργό τρόπο, ιδιαίτερα στη σύγκρουση στο Άνω Καραμπά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν συστηματικά απούσα θα έλεγα όλα αυτά τα χρόνια και τώρα θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας διεθνής διαιτητής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός από τις δύο εμπλεκόμενες ε, ε, πλευρές. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει συμφιλιωτικά προγράμματα, επαφές ανάμεσα στους πληθυσμούς και στους λαούς της περιοχής. Οι συγκρούσεις στην περιοχή θα βοηθήσουν και τον επαναπατρισμό εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα μέσα και την εμπειρία να δημιουργήσει μια πιο ανεκτική ατμόσφαιρα στο Νότιο Κάφκασο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και τη δική της ιστορική εμπειρία και να δείξει στους λαούς της περιοχής ότι μπορεί να συμβιώσουν εν ειρήνη και ευημερία. Είναι βασικός στόχος της Ένωσης να πείσει τους ηγέτες και τους λαούς της περιοχής, τις ψυχές και τις καρδιές των ανθρώπων της περιοχής, ότι η περιοχή τους θα μεγαλώσει και θα αναπτυχθεί με εμπιστοσύνη και συνεργασία. Ο Επίτροπος Φίλε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές Κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ ευτυχής που συμμετέχω εδώ σε αυτήν την ε, συνεδρίαση που αφορά τον Νότιο Κάφκασα. Ήδη είχαμε καλή συζήτηση για τον Νότιο Κάφκασο με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στις 28 Απριλίου, λίγο μετά την επίσκεψή μου στην περιοχή. Εργάζομαι από αυτή τη έκθεση. Ε, θεωρώ πω είναι μια πολύτιμη συμβολή στον προβληματισμό για το πώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να οικοδομήσει μια ισχυρότερη ε, σχέση με την Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν και την Γεωργία. Θα πρέπει να σας θυμίσω πως έχουμε ένα στέρεο πλαίσιο δέσμευσης με την ε, παγιωμένη ευρωπαϊκή πολιτική γυτνίαση και την ανατολική εταιρική σχέση που ξεκίνησε πέρσι. Με μεγάλες προτεραιότητες όσον αφορά τις εξωτερικές μας σχέσεις, ε, η επιτυχής υλοποίηση της, ε, εταιρικής, της ανατολικής εταιρικής σχέσης θα ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις μας με τους εταίρους αυτούς. Να υπογραμμίσω τα εξή. Την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν δημοσίευσε την πρώτη έκθεση πρόοδου για τις χώρες του Νότιου Καυκάσου το πρόγραμμα δράσης και την ε, τακτική αξιολόγηση της εφαρμογής των προγραμμάτων παραμένουν ένα βασικό εργαλείο για τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές καθώς και για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη φορά ε, επιλέξαμε μία αξιολόγηση για τις χώρες του Νότιου Καυκάσου. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα πορίσματα στη βάση για επεκτεταμένες ε, ε, διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη, με εσάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τους εταίρους μας στην περιοχή, ώστε να έχουμε τη δική τους ανταπόκριση, το feedback, αν έχουμε τα σωστά εργαλεία και μέσα, αν ε, τα ποσά τα οποία οι πόροι που έχουμε στη θέση μας είναι κατάλληλοι, καθώς και αν η ταχύτητά μας και οι προσπάθειές μας κατευθύνονται την σωστή κατεύθυνση. Ε, θα πρέπει η πολιτική μας να είναι πιο συνεκτική και να οδηγηθούμε σε υψηλότερο βαθμό συμμετοχή των γειτόνων μας. Θα είναι και εξαιρετική περίπτωση ώστε να υποστηρίξουμε την παροχή κατάλληλων πόρων μέσω των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα δόθη έγκριση από το Συμβούλιο για την έναρξη ε, συμφωνιών σύνδεσης με την Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν και την ε, Γεωργία. Αυτό είναι ένα σαφέ μήνυμα της ε, στεναρής μα δέσμευση για συνεργασία ανάμεσα στην Ένωση και τις χώρες του Νοτιού Καυκάσου επί τη βάση κοινών αξιών και αρχών, ε, δημοκρατία, κράτος δικαίου και σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κομισιόν ήδη προετοιμάζεται για την εκκίνηση τέτοιων διαπραγματεύσεων που αναμένεται να γίνει στις επόμενους μήνες. αυτοί οι δύο τομείς ε, αποδεικνύουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει μια συνολική παγιωμένη πολιτική για τις χώρες του Νοτιού Καυκάζου και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη στρατηγική πλήρως ώστε αυτή η περιοχή να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος ε, έκανε μια πολύ σημαντική ε, έκθεση την οποία, την οποία εκτιμούμε ιδιαίτερα και ε, οι απόψεις μας συγκλίνουν σε πολλά θέματα. Η σταθερότητα και η ασφάλεια του Νότιου Καυκάζου έχει άμεσο αντίκτυπο στην Ένωση, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται την ευθύνη για υποστήριξη της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν συνδέσεις μεταφορές και υποδομές. Η στήριξη του κράτους δικαίου θα βοηθήσει το εμπόριο και τις επενδύσεις καθώς και την κινητικότητα των ανθρώπων και οι ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες σύνδεσης θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο σωστό δρόμο όσον αφορά τις σχέσεις με την Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν και την Γεωργία. Είμαστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός επικοδομητικού πλαισίου και πρόκειται για κοινή προσπάθεια. Η δέσμευση των εταίρων μας του Νοτιού Καυκάσου για προσέγγιση προς την Ευρώπη θα πρέπει να μεταφραστεί σε περαιτέρω πρόοδο προς τη δημοκρατία, την οικονομία της αγοράς και την πολιτική σταθερότητα. Ας καλέσουμε την Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν και την Γεωργία να προχωρήσουν στις προσπάθειές τους για ε, μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία που θα είναι σε ειρηνικέ σχέσεις με τους γειτονές της. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εξ Κομισιόν, εξ της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Καζάκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο συντονιστής της ΣΑΛΤΕ. Θα ήθελα να τονίσω την θέση τη Επιτροπή μα ότι είναι απαραίτητη μια στρατηγική για τον Νότιο Κάφκασο. Είναι ιδιαίτερα λεπτή αυτή η έκθεση γιατί αυτή η στατιστική είναι κεφαλαιώδης για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας πλήρως την πολιτική γειτονία και να τονίσουμε το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω ενό γενικού μεσαισιαγωγικά παίκτη για την ασφάλεια τη περιοχή. Υπάρχουν πολλέ δυνατότητε στον τομέα τη ενέργεια, τη ευκυβερνησία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θεσπίσει στόχους οι οποίοι είναι στόχοι προτεραιότητος. Θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση γεωστρατηγικού χαρακτήρα της Αρμενίας του Αζερβαϊτζάν, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της Ρωσίας είναι απαραίτητο να εξαλείψουμε και όλους τους εμπορικούς φραγμούς για να μπορέσουμε να δώσουμε και μια μεγαλύτερη τόνωση στις εμπορικές ανταλλαγές, κάτι το οποίο θα επιτρέψει να συμβάλλουμε περισσότερο στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη σταθερότητα της σύνολης περιοχής. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιζητήσει τη δημιουργία μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών στον Κάφκασο, διότι με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλει στο να ρυθμιστούν οι υποβόσκουσες συγκρούσεις και επίσης θα ευνοήσει την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας των χωρών της περιοχής και ζητώ από την Κομισιόν να αναλάβει να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ κύριε Καζάκ. Από τις πολιτικές ομάδες συνεχίζουν ομιλητές. Στις 12 πρέπει να ψηφίσουμε όμως. Γι' αυτό σας παρακαλώ να παραμείνετε στα πλαίσια του χρόνου σας. Δύο λεπτά για, από την ομάδα του ΕΛΚ, την κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ψηφίσουμε πράγματι για την έκθεση για την στρατηγική της Ένωσης για τον Νότιο Κάυκασο. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει πιο ενεργό ρόλο σε αυτή την περιοχή. Ως και συγκήτρια εγώ για το ΕΛΚ έχω εργαστεί πάρα πολύ σκληρά για να τονίσω το ρόλο της Ένωσης στο Νότιο Κάυκασο και για το τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε πρακτικά τις ε, χώρες εκείνες και να τις φέρουμε πιο κοντά στην Ένωση. Κάθε μία από αυτές τις χώρες, σύμφωνα με τις ε, δικές της ε, ιδιαιτερότητες, θα κινηθεί. Αναφέρουμε λοιπόν κάποια πράγματα στην, στρατηγική, στην έκθεση για το πώς θα πραγματοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Πρέπει πρώτα να αυξηθεί ο ρυθμός των ε, σχετικών ε, συνομιλιών για να οδηγηθούμε σε μια περιοχή ελευθερου εμπορίου με τον ε, Νότιο Κάφκασο. Όλες οι χώρε περιοχή, Αρμενία, Γεωργία, Αζερβαϊτζάν ήταν δημοκρατίε τη Σοβιετική Ένωσης, οπότε η Ρωσία ασκεί ακόμα μεγάλη επιρροή στην περιοχή. Επίση για να υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια και ελευθερία, πρέπει να έρθει πιο κοντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή από ό,τι είμαστε αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευρωπαϊκή προοπτική για αυτές τις χώρες και είναι σημαντικό η Ένωση να αντιληφθεί την κατάσταση εκεί πέρα και την ευθύνη της. Γνωρίζω επίσης πως πρέπει να έχουμε κατά νου τις μακροχρόνιες συμβούσεις σε αυτή την περιοχή και το τι μπορεί να γίνει για να αποτραπούν. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη για το ότι στο κείμενο αυτό επανειλημμένα τονίζουμε την άνεφόρον στήριξή μας για το σεβασμό των συνόρων και των δικαιωμάτων στην περιοχή και πρέπει να αναγνωρίσουμε και την, ε, να απορρίψουμε τη ρωσική αναγνώριση της Νότιας Οσετίας και της ε, Απχαζίας. Οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω να στηρίξετε τις τροπολογίες ε, ΕΛΚ Σοσιαλδημοκρατών και Πρασίνων. Σας ευχαριστώ για δύο λεπτά για τους σοσιαλιστές ο κύριος Φόποντα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρα, πρώτα απ' όλα ευχαριστήσω τον κύριο Κύριλοφ για την εργασία του, την ευρύτατη, που αποτελεί μεγάλη συνεισφορά για τη στρατηγική μας στην περιοχή. Ε, εγώ βρέθηκα πρόσφατα στην ε, Τυφλίδα και φαίνεται πως ε, λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα πως η περιφερειακή συνεργασία είναι κάτι που μας το επιβάλλει η Ευρώπη και αυτό δείχνει την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη. Γιατί λένε πως θέμε να συνεργαστούμε αλλά ίσως να μην έχουμε και άλλη λύση αν μας το επιβάλλει η Ευρώπη. Κοιτάξτε, για εμάς στην Ευρώπη αυτό αποτελεί την βάση της ειρηνική εξέλιξη της συνεργασίας και το ίδιο πρέπει να γίνει και στο Νότιο Κάφκασο. Και βεβαίω υπάρχει εκεί πέρα η πίεση του πρώην μεγαλοδερφού της ε, μεγάλη δύναμη της Ρωσίας και δεν ξέρουμε τι επίθεση θα έχει αυτό για τη συνεργασία αυτών των χωρών βεβαίως. Αυτό αφορά και τις ε, χώρες εκεί τις ε, γειτονικέ και εδώ πέρα αναφέρομαι στην Τουρκία με την οποία συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και εγώ θα επιθυμούσα τα προβλήματα αυτά στα οποία είναι συνυπεύθυνη η Τουρκία ή θα μπορούσε να έχει μια ε, συνυπευθυνότητα, δηλαδή τα προβλήματα με την γειτονική χώρα, την Αρμενία και το ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ να λυθούν ως πακέτο. Δεν υπάρχει νομίζω κανένα πρόβλημα να φύγουν τα αρμενικά στρατεύματα εκτός των περιοχών του Ναγκόρνο Καραμπάχ για να δημιουργηθούν επίσης και καλύτερες σχέσεις μεταξύ Αρμενίας και Τουρκίας. Εμείς στην ομάδα μας λέγαμε πάντα πως πρέπει να υπάρχει αυτή η Ένωση, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Μαύρης και νομίζω αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και για τους γείτονες εκεί πέρα, την ε, Τουρκία, τη Ρωσία. Και νομίζω πως θα μπορούσε να βρεθεί μια τέτοια συνέχεια μέσω αυτής τη Ένωσης, η οποία αυτή τη στιγμή αποτελεί όραμα, αλλά μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ για τους φιλελεύθερους δημοκράτες. Δυόμιση λεπτά η κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σαν σκιώδη συζητήτρια για τους φιλελευθέρους θα ήθελα να πω ότι η έκθεση αυτή είναι μια εξαιρετική βάση για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της περιοχής του Νοτιού Καυκάσου. Είναι μια έκθεση η οποία σαφώς και προσφέρει προστιθέμενη αξία στις γνώσεις μας για την περιοχή και ευχαριστώ τον κύριο Κυριλόφ για την εξαιρετική δουλειά την οποία έχει κάνει και τη συνεργασία, με τη συνεργασία των υπολείπων πολιτικών ομάδων νομίζω ότι το 2010 μπορεί να είναι μια ακομβική στιγμή ευκαιρίας για την περιοχή αυτή. Τα τρία προβλήματα της περιοχής, Αυχαζία, Οσετία και ε, Βόρειο Καραμπάχ, ε, μπορεί να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη ψυχραιμία και αποτελεσματικό τρόπο. Η ευρωπαϊκή διπλωματία μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση σε κάποια από τα προβλήματα αυτά. Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης και το πολύ σημαντικό θέμα για μας, το της ε, ασφάλειας στον τομέα της ενέργειας. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξομαλύνουμε τις ε, εντάσεις, τις αιστείες εντάσεως που υπάρχουν στην περιοχή αυτή και θα πρέπει ταυτόχρονα να ολοκληρώσουμε τις προσπάθειες που έχουμε ήδη ξεκινήσει για τον εκδημοκρατισμό των χωρών της περιοχής. Ε, υπάρχουν βέβαια στην περιοχή αυτή κάποιες προκλήσεις ολοκληρωτισμού και υπάρχουν δημοκρατικά ελλείμματα και θα πρέπει να υπερκεραστούν. Μέσω των προγραμμάτων μας θα πρέπει να οδηγήσουμε σε αηφόρες μορφές ανάπτυξης, κάτι το πολύ σημαντικό για τη συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να βοηθήσουμε να ξεπεραστούν οι νοοτροπίες που οδηγούν στην διαφθορά και στις συγκρούσεις. Για να το πετύχουμε αυτό απαιτείται να γίνεται σεβαστή η βούληση των λαών της περιοχής από τις κυβερνήσεις. Η έκθεση τα υπογραμμίζει με σωστό τρόπο όλα αυτά και αναφέρεται και σε επιμέρους σημεία τα οποία έχουν σημασία για μας όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, και νομίζω ότι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα μεμονωμένα κράτη-μέλη μια στρατηγική σχέση με τις χώρες αυτές ε, είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ για την ομάδα των Πρασίνων και για δύο λεπτά η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα όπως και οι προλαλήσαντες να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Κυρίλοφ για την πολύ καλή συνεργασία που είχε με όλους τους κοιόδες συζητητές και για την πολύ καλή ποιότητα αυτής της έκθεσης, η οποία είναι μια πλήρης και περιεκτική έκθεση. Θέλω να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία και μόνο τα οποία δεν αντανακλώνται ιδιαίτερα στην έκθεση, αλλά μου φαίνονται πάρα πολύ σημαντικά. Οι τρει αυτές παγωμένε σειράξεις που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εμπόδιο για να μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία αλλά και στις ίδιες τις χώρες αποτελεί ένα πραγματικό εμπόδιο στην ανάπτυξή τους. Αν έχει κανείς ένα εξωτερικό εχθρό πραγματικό ή φανταστικό, τότε αυτό εμποδίζει το να αναλάβει την ευθύνη να κάνει τα απαραίτητα μέσα στην ίδια του τη χώρα και αποτελεί πολλές φορές ένα πρόσημο για να μην πράξει τέτοια πράγματα. Το να μπορέσουν λοιπόν να φύγουν οι πολιτικές των χωρών αυτών από στρατηγική οτικές δραστηριότητες και δαπάνες οι οποίες έχουν ανέβει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και να δοθούν προς το αντιμετώπιση κοινωνικών, περιβαλλοντικών ή οικονομικών προβλημάτων του πληθυσμού είναι κάτι το απαραίτητο και αυτά τα αναφέρει η έκθεση του κυρίου Κυρίλοφ. Επίσης, σε ό,τι αφορά την σύγκρουση μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας, φάνηκε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αφοπλισμό όχι μόνο σε επίπεδο όπλων, αλλά και σε επίπεδο ρητορική, εναντίον μια γλώσσα η οποία είναι παραπλανητική και δημογωγικού χαρακτήρα. Είναι απαραίτητο οι χώρε αυτέ να προχωρήσουν σε ένα επίπεδο δημιουργία συνθήκων ειρήνη. Και επίση είναι απαραίτητο να υπάρξει μεγαλύτερη δημοκρατικοποίηση, υποστήριξη τη κοινωνία των πολιτών, προστασία θρησκευτικών, εθνοτικών, σεξουαλικών μειονοτήτων. Στο Παραδείγματο χάρη στο Αζερβαϊτζάν, δύο νέοι ε, στο ίντερνετ, οι οποίοι τόλμησαν να επικρίνουν την κυβέρνηση, του στείλαν για δύο χρόνια στι φυλακέ. Είναι απαραίτητο επίση να υποστηρίξουμε την ελευθερία των μέσων, που είναι πρόβλημα σε όλε αυτέ τι χώρε. Όλα αυτά είναι πτυχέ οι οποίε αναφέρονται στην έκθεση αυτή, αλλά όπω είπε και ο... η πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο την περιφερειακή διάσταση αλλά και την υπερμεθοριακή διάσταση και περιμένουμε από την Κομισιόν να λάβει πλήρω υπόψη αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ από τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστές. Για δύο λεπτά ο κύριος Κύριε Πρόεδρε, όπως κάνει σαφές η έκθεση, κύριε Ρίλοφ, οι χώρες του Νότιου Καυκάσου είναι σημαντικές στρατηγικές για την, ε, στρατηγικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ενέργεια, δηλαδή φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τον Νότιο Καύκασο και διαμετακόμιση ε, ενέργειας μέσω αυτής τη περιοχής, αλλά και για στρατηγικού λόγους. Δυστυχώ, παραμένουν οι παγωμένε σειράξει σε αυτή την περιοχή. Κύριο λόγο για, γι' αυτό είναι η αναγνώριση κατά την άποψή μα η αναγνώριση της Απχασίας και της Νότιας Οσετίας από τη Ρωσία και η εισβολή στο κυρίαρχο έδαφος της ε, Γεωργίας. Οι μηχανισμοί της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας θα πρέπει να λειτουργήσουν για να ανταμείψουμε τις προσπάθειες της Γεωργίας να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες της για προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται λοιπόν να προχωρήσουμε και σε μέτρα ε, σύνδεση με τι χώρε αυτέ, με φιλελευθερωποίηση των καθεστώ προξενικών ε, θεωρήσεων κτλ. Και ω φίλο τη Αρμενία θεωρώ ότι η τελική μορφή αυτή τη έκθεση είναι πιο ισορροπημένη από την αρχική. Εξακολουθώ όμω να ανησυχώ για ορισμένε διατάξει στην έκθεση αυτή που φαίνεται να αντιβαίνουν στην επίσημη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την επίλυση του προβλήματο του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η Αρμενία έχει κάνει θαραλές προσπάθειες για να ξεπεράσει το αδιέξοδο για το Ναγκόνο Καραμπάχ. Επίσης έχει επιζητήσει μια ομαλοποίηση των σχέσεων της με την Τουρκία, κάτι το οποίο θα σταθροποιήσει περισσότερο το Νότιο Κάφκασο, εφόσον βέβαια και η Τουρκία επικοδομητικά και χωρίς προϋποθέσεις ανταποκριθεί σε αυτή την πρωτοβουλία. Αν ανοίξουν λοιπόν τα σύνορα αυτά, αυτό όχι μονάχα θα το εμπάργο για την Αρμενία που την έχει ταλανίσει επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα επιτρέψει όμως η οικονομική ευμάρεια στις ε, υπανάπτυκτε περιοχέ τη Ανατολική Τουρκία. Υπάρχει και συμφέρον λοιπόν για την Τουρκία να προχωρήσει προ αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Τουρκία μπορεί να διατηρεί αενάω κλειστά τα, τα, τα σύνορά τη με την Αρμενία λόγω τη λεγόμενη αλληλεγγύη τη με το Αζερβαϊτζάν σε σχέση με τη σύραξη του Ναγκόρνο Καραμπάχ θα ήταν σαν η Ελλάδα να έκλεινε τα σύνορά της στον Εύρο στην Κύπρο για λόγους αλληλεγγύης με τους Κύπριους μετά από την κατοχή της Βόρειας Κύπρου. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουμε στο ελεύθερο εμπόριο και τα ανοιχτά σύνορα που είναι απαράγραπτη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ειρήνη στην περιοχή μας και στο Νότιο Κάφκασο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνο και την Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Ένα λεπτό κύριο Προβέρα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Λόφ ο τομέας τον οποίο ανέλαβε είναι ένας τομέας γεμάτος δυσκολία αλλά γεμάτος ευκαιρίες επίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει ένα ενδιαφέρον σχέδιο εταιρικής σχέσης με τις χώρες αυτές και έχει συμφωνηθεί σε ένα πρώτο επίπεδο με το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία και τη Γεωργία. Απαιτούνται όμως περαιτέρω μέτρα και προσπάθειες στον τομέα της ενέργειας, της οικονομίας, της πολιτικής αλλά και στον τομέα της ασφάλειας για να αντιμετωπιστούν οι εντάσεις ανάμεσα στην Τουρκία, την Αρμενία και τα προβλήματα της Οσετίας και του Νακόρνο Καραμπά. Ένα τέτοιο σχέδιο σαν αυτό που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν πολύ πιο αποδοτικό εφόσον οι τρεις αυτές χώρες σεβαστούν αμοιβαία την εδαφική τους κυριαρχία και ακεραιότητα και θέσουν τις βάσεις ε, για την επίλυση των προβλημάτων που παραμένουν χαίνοντας την περιοχή. Θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι εδώ θα πρέπει όλες οι χώρες να αναγνωρίσουν το απαραβίαστο των εξωτερικών συνόρων των χωρών αυτών, κάτι το οποίο πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που δεν θα πρέπει να αλλάξουν ποτέ με χρήση στρατιωτικής βίας. Για ένα λεπτό για τους άγραφτους βουλευτές, ο Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω πρώτα απ' όλα κυρίες και κύριοι πως οι κύριοι Κύριλοφ και Καζάκ ανήκουν σε πολιτικά κόμματα τα οποία συστηματικά ψηφίζουν στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο κατά της αναγνώρισης της αρμενικής γενοκτονίας. Οπότε είναι περίεργο το ότι αναφέρονται διαφορετικά πράγματα σε αυτή την έκθεση, όπως είπε ο κ. Τζανάκα. Παραδείγματο χάρη για τον Αγκόρνο Καραμπάχ ήρθαν σε επαφή μαζί μου κάποιες οργανώσεις και μου είπαν ε, πως ε, η έκθεση αυτή δεν ε, σέβεται τα κριτήρια της Μαδρίτης ούτε ήρθαν σε συνεννόηση με την ομάδα του Μίνσκ. Αυτή είναι λοιπόν η επικοδομητική μου κριτική προς τον συνάδελφο τον κύριο Κυρίλοφ γιατί νομίζω πως η μονομερής θέση υπέρ μίας μονοπλευράς δεν θα λύσει τη σύγκρουση. Χρειαζόμαστε μια ευέλικτη θέση που θα αντικατοπτρίζει όλες απόψεις γιατί αλλιώς δεν θα λυθεί ποτέ η σύγκρουση. Ευχαριστώ κύριε Στογιάνοφ. Περνάμε στους ε, λοιπούς ε, ομιλητές για 1,5 λεπτό ο κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θεωρώ πως ο εκδημοκρατισμός, η ορθή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πράγματα στα οποία πρέπει να εδρεωθούν η σχέση μας με τις χώρες αυτές. Γι' αυτό η συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο θα αυξήσει και το δυναμικό συνεργασίας αυτών των χωρών με την Ένωση. Πολλές από τις διαστάσεις οικονομικής συνεργασίας είναι επίσης σημαντικές. Να τονίσω κάποιες όπως παραδείγματο χάρη η ενεργειακή ασφάλεια, ειδικά όταν μιλάμε για τόσα έργα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ο Αγώνα Ναμπούκο. Η Κασπία και η Μαύρη Θάλασσα έχουν ζωτική σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης και η στρατηγική της Ένωσης σωστά αναγνωρίζει αυτά τα στοιχεία. Τρία συγκεκριμένα στοιχεία θα ήθελα να τονίσω σύντομα. Ένα από αυτά είναι η ανάμειξη των τοπικών αρχών στη διασυνοριακή συνεργασία γιατί χρειαζόμαστε και ισχυρή τοπική συνεργασία. Μετά έχουμε το θέμα του ένταξη του Αζερβαϊτζάν στον ΠΟΕ και πρέπει να βοηθήσει να δώσει τεχνική αρρωγή κομισιών στο Αζερβαϊτζάν και τρίτον και τελευταίον τεχνική αρρωγή για ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος ε, και του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο Νότιο Κάφκασο έτσι ώστε οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές να έχουν καλύτερες προοπτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βίνκλερ. Ο κύριος Σεβερίν για δύο λεπτά έχει το λόγο. Κύριε αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση Κυρίλοφ αναφέρεται στην ανάγκη να υπάρξει μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Κάφκασο και πιστεύω πράγματι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια τέτοια στρατηγική. De facto αυτή η στρατηγική χρειάζεται στόχους και οι στόχοι προϋποθέτουν μια γεωστρατηγική ταυτότητα. Θα πρέπει να βρούμε τη γεωστρατηγική μας όμως ταυτότητα για να μπορέσουμε να ξέρουμε ποια ακριβώς είναι αυτή η ταυτότητα. Τι επιζητούμε στο Νότιο Κάφκασο. Σταθερότητα, ανοιχτό χαρακτήρα της περιοχής και διαλειτουργικότητα. Μια πολιτική δημοκρατία, μια δημοκρατία σταθερή στην περιοχή αυτή. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει αυτή την περιοχή μέσα στην εταιρική σχέση της Ευρώπης με την Ανατολική Ευρώπη είναι το γεγονό ότι όλε αυτέ οι χώρε έχουν και τη δική του ιδιαιτερότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί δέοντα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και το ρόλο τη Τουρκία στην περιοχή αυτή <clears throat> και να χρησιμοποιήσουμε τι διαπραγματεύσει μα με την Τουρκία ω ένα πλαίσιο για να αναπτύξουμε περισσότερο μια εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία για να αντιμετωπίσουμε τοπικέ και περιφερειακέ προκλήσει στην περιοχή. Όπω τονίστηκε, η Τουρκία μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επίση ότι αυτή η περιοχή είναι τμήμα τη κοινή γειτονία μα με τη Ρωσία και θα πρέπει να βρούμε τρόπου να προωθήσουμε κοινέ πολιτικέ σε αυτή την κοινή γειτονιά. Τα θέματα ασφάλεια καταρχήν πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επίση θέματα ενέργεια. Όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τριμερεί συζητήσει και διαπραγματεύσει. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να μα βοηθήσει να προωθήσουμε λύσει για τι τοπικέ, όπω αναφέρονται, παγωμένε σειράξει. Θα πρέπει να δεχτούμε όμως ότι αυτές οι συγκρούσεις, οι σειράξεις είναι τμήματα ενός ευρύτερου καμβά που έχει μεγαλύτερη σημασία και σε γενικότερο επίπεδο. Επομένω, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως τμήματα ενός πακέτου. Πρέπει επίσης να ξεπεράσουμε τις αμφισημίες και να κατανοήσουμε ότι οι αρχές της αυτοδιάθεσης και της εδαφικής ακεραιότητας δεν μπορούν πάντα να συμβαδίζουν. Και τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε να διοργανώσουμε μια διάσκεψη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στο Νότιο Κάφκασο, ώστε να υπάρξει μια συμφωνία σταθερότητα για την περιοχή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σεβερίν. Ένα λεπτό. Ο κύριος Πορέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ήτροπε. Σαν εκπρόσωπος γενικότερα της Αρμενίας θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη για μια συνεκτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Στήριξη της ελευθερίας, στήριξη των δικαιωμάτων των ε, πολιτών, στήριξη της δημοκρατίας, στήριξη της ελεύθερης αγοράς. Γι' αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία που θα οδηγήσει ε, σε εταιρική σχέση με την Αρμενία και θα βοηθήσει η συνεργασία αυτή την ε, Αρμενία να ξεκινήσει ουσιαστικότερες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της πολιτικής και της οικονομίας και η Γεωργία έχει προχωρήσει, ε, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον σε επιχειρηματικό επίπεδο. Είναι ε, στην ένατη θέση στην περιοχή αυτή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκτιμήσει το γεγονός ότι ο πρόεδρος Σαχασβίλη εφαρμόζει ένα σωστό παράδειγμα και για τις άλλες χώρες. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, στις 9 Μαΐου εδώ με τον ε, κύριο Μπούζεκ εορτάσαμε την 60η επέτειο της ε, δήλωσης Σουμάν με 20.000 άτομα και η εναλλακτική λύση είναι ο Νότιος Κάυκασος. Είτε θα έχουμε ένα τέτοιο τέτοια φαινόμενα σε παγκόσμια κλίμακα όπως είχαμε στον Μεσοπόλεμο ή θα έχουμε εξέλιξη όπως στην Ευρωπαϊκή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και δίκιο έχει και ο κύριος Κυρίλοφ και ο κύριος Φόποντα πως εάν συνεργαστούν αυτές οι τρεις χώρες θα μπορέσει να μειωθεί και η εξωτερική επιρροή και η ρωσική επιρροή. Οπότε υποστηρίζω την Αρμενία στις ε, προσπάθειες της αναγνώρισης ε, της ε, γενοκτονίας από τους Οθωμανούς, αλλά θα ήταν και πιο αξιόπιστη αν απέσυρε τα στρατεύματά της από το Αζερβαϊτζάν και χρειαζόμαστε επιγόντως λύση και για το Καραμπάχ και για τις κατεχόμενες αζερικές περιοχές και μια σταθεροποίηση της γεωργίας γιατί αυτή τη στιγμή εάν διαλυθεί όπως θέλουν κάποιοι στη Μόσχα θα αποσταθεροποιηθεί ολόκληρη η περιοχή. Γι' αυτό αυτές είναι, αυτά είναι τα σημαντικότερα ζητήματα. Ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει, ζήτημα των, τα ζητήματα των μειονοτήτων και βεβαίως να επανέλθουν στις αιστείες του οι εκδιωγμένοι. Δεν είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα να μιλάμε για διώξεις και εκτοπισμούς. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο ευαίσθητοι και δραστήριοι. Για δύο λεπτά. Παλέκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον συνάδελφο Κυρίλοφ για την τόσο σωστά ε, διατυπωμένη και προσεκτικά συνταγμένη εκθεσή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και την Αρμενία να κάνουν όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να μπορέσουν να αναπτυχθούν ως δημοκρατικά σύγχρονα κράτη. Αυτό σημαίνει να υπάρχει και σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και σεβασμό των θέσεων τη αντιπολίτευση στι χώρε αυτέ. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να υπάρχει περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή αυτή και τα τρία αυτά κράτη του Νοτίου Κάφκασου έχουν <clears throat> αντιμετωπίσει πρόσφατα συγκρούσεις παγωμένες ή μη. Και μέσα στην ε, αντιπαράθεση αυτή που έχει γίνει, είναι, φανερό ότι η μόνη λύση για το μέλλον είναι να, υπάρξουν συνεργασία, να υπάρξει συνεργασία και διαπραγματεύσει και όχι να είναι στραμμένο το βλέμμα του μονάχα προ το παρελθόν. Οι χώρε αυτέ θα μπορέσουν να αυξήσουν τη δυνατότητά του να έχουν μια προοπτική ευρωπαϊκού χαρακτήρα όταν μπορέσουν να συνεργαστούν και μεταξύ του. Αυτό όμω σημαίνει ότι θα πρέπει εμεί να κάνουμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τι χώρε αυτέ που έχουν αυτή τη στιγμή υστερήσει σε διάφορα επίπεδα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο στην περιοχή αυτή, ιδίω στα προγράμματα καταπολέμηση τη ένδυα, η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, ανδρών και γυναικών, να υπάρξει μεγαλύτερη επένδυση στην υγεία και στην εκπαίδευση και θα πρέπει να καταβάλουμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να υπάρξει μια άμεση επαφή μεταξύ των πολιτών των χωρών του Νοτιού Καυκάσου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των φοιτητών που εμπλέκονται σε προγράμματα ανταλλαγών και κινητικότητα. Όλο αυτό είναι και προ το δικό μα συμφέρον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παλέτσκι. Για ένα λεπτό κύριο Τσαρνέσκι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, βρισκόμαστε ενώπιον ενό πολύ σημαντικού βήματο προ τα εμπρό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή μπορεί να ανοίξει την πόρτα στι χώρε του Νοτιού Καυκάσου που έχουν ένα σαφή ευρωπαϊκό χαρακτήρα, τη Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Αλλά αυτό το βήμα έρχεται κατόπιν εορτής. Είναι κρίμα ότι εμείς δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, να πράξουμε αυτά που πράττουμε σήμερα πριν από δύο χρόνια, τότε που έγινε η επέμβαση της Ρωσίας στην Γεωργία. Παρ' όλα αυτά είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση και η ελπίδα μου είναι ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε το σωστό πολιτικό περιεχόμενο σε αυτή την πρωτοβουλία. Ελπίζω ότι η κοινοβουλευτική συνέλευση Euronest θα είναι ένα ε, αποτελεσματικό εργαλείο για να υποστηρίξει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες αυτές. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι θα έπρεπε κάποιοι από εμά να μιλήσουν με στεντόρια φωνή για τη δημοκρατία στον μεγάλο γείτονα και αδελφό των χωρών αυτών, τη Ρωσία. Δεν πρέπει να έχουμε δύο μετά και δύο σταθμά. Ενάμιση λεπτό. Ο κύριος Λίεσεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν και η Γεωργία είναι ευρωπαϊκές χώρες και ευρωπαϊκά έθνη. Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και εταίροι σε πάρα πολλές διεθνείς συμβάσεις, συμφωνίες και σχέδια συνεργασίας μεταξύ των οποίων και η εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα κάθε χώρα στην αυτοδιάθεση και στην διαμόρφωση του μέλλοντος του. Θα πρέπει να μην κολλάμε σε αρχαϊκές επιρροές, σε αρχαϊκές αντιλήψεις περιζώνων επιρροής. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την εδαφική ακαιρεότητα της Γεωργίας και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να διατηρηθεί η ακαιρεότητα αυτή και θα πρέπει η Ένωση να θεωρηθεί σαν εγγυήτρια ασφάλειας για την περιοχή. Δυστυχώς όμως κάποια τμήματα της συμφωνίας του Σεπτεμβρίου του 2008 δεν εφαρμόζονται. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στη Γενέβη και ίσως τις διμερείς επαφές μας με τις ε, ρωσικές αρχές, τις αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας να εμείνουμε λίγο περισσότερο. Σχετικά με τις θεωρήσεις και τις νέες ρυθμίσεις θεωρήσεων. πρέπει να βοηθήσουμε τους πληθυσμούς της περιοχής να έρχονται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αφορά και τις τρεις χώρες. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Κούτας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε δεδομένης ε, της ε, σημασίας της γεωπολιτικής κατάστασης της Αρμενίας, Αζερβαϊτζάν και της Γεωργίας σε σχέση με την Ένωση την Τουρκία, τη Ρωσία και το Ιράν, χρειαζόμαστε μια στρατηγική για τον Νότιο Κάφκασο η οποία θα βασίζεται στην οικονομική ανάπτυξη και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το εμπόριο είναι ένα από τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει και συμφωνίες ελευθερου εμπορίου με αυτές τις χώρες που θα δώσουν όθηση στις ε, ξένες επενδύσεις ε, και θα προωθήσουν την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Επίσης η ενεργειακή ασφάλεια είναι μια βασική, ένα βασικό μέλημά μας σε αυτή την περιοχή και πρέπει βεβαίως να ολοκληρωθούν και οι διαπραγματεύσεις για τον Αμπούκο και να υποστηρίξουμε τα έργα ενεργειακής αποδοτικότητας και εναλλακτικών πηγών ενέργειας στον Νότιο Κάφκασο. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο Σκόβαλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Γεωργία και η Αρμενία και σύμφωνα με την άποψη των συντακτών της έκθεσης εφαρμόζουν ε, κατ' ουσίαν τη στρατηγική γειτονία με την Ένωση. να το λάβουμε αυτό υπόψη, όπως και να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητε της κάθε χώρα. το ε, τομεί όπως ε, ο πολιτισμό, οι μεταφορές, η προστασία του περιβάλλοντος. Συχνά όταν μιλάμε λοιπόν για αυτέ τις περιοχές μιλάμε για παγωμένες συγκρούσεις, εθνοτικά προβλήματα και είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Αλλά για να απαντήσουμε στα προβλήματα αυτής της περιοχής πρέπει να στηρίξουμε τον εξυγχρονισμό αυτής της περιοχής έτσι ώστε να μην ε, παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο οι συγκρούσεις. Συχνά φαίνεται να ξεχνάμε πως η Γεωργία μόλις βγήκε από έναν πόλεμο. Για να μην έχουμε λοιπόν άλλους πολέμους σε αυτήν την περιοχή πρέπει να υποστηρίξουμε τον εξυγχρονισμό γιατί η Γεωργία, το Αζερβαϊτζάν και η Αρμενία έχουν ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και πρέπει να τη στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ για 1,5 λεπτό ο κύριος Κόβατσεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην μιλήσω με μεγάλη ταχύτητα. Εγώ υποστηρίζω την έκθεση του κυρίου Κύριλοφ, ο οποίος τονίζει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή αυτή. Η ανάπτυξη του Νοτιού Καυκάσου θα βοηθήσει και τη συνεργασία στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν έχει ακόμα μια σαφή στρατηγική. Ελπίζω θα το συζητήσουμε όσον ούπο το θέμα αυτό. Θέλω να τονίσω επίση και τι ανησυχίε μου για την βραδιπορία της διαδικασίας κύρωση των πρωτοκόλων που υπογράφηκαν τον προηγούμενο Οκτώβριο μεταξύ Τουρκία και Αρμενία. Νομίζω ότι καμία από τι δύο χώρε δεν θα πρέπει να θέσει προποθέσει για την κύρωση αυτών των πρωτοκόλων. Γιατί έχουν μεγάλη σημασία και για του δύο λαού. Οι διαπραγματεύσει για το άνοιγμα των συνόρων και τι διπλωματικέ σχέσει μεταξύ των δύο χωρών έχουν πολύ μεγάλη σημασία και επίση φυσικά το ζήτημα του Ναγκόνο Καραμπάχ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χωριστά από τα θέματα αυτά. Και η Τουρκία αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν ένα πιο σημαντικό ρόλο στην επίλυση του θέματο του Ναγκόνο Καραμπάχ. Έχουμε εμπειρία από τα Βαλκάνια. Πιστεύω ότι έχουμε και εμπειρίε από την Γεωργία. Γι' αυτό νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή θέση για να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή αυτή. Ένα ευμαρή Νότιο Κάφκασο είναι προ το συμφέρον όλων μα και θα πρέπει να υπομισθούμε και τις ευθύνες μας για κάτι τέτοιο. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε ένα ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα μπορέσει να αποτελέσει τμήμα της ομάδας του Μίνσκ και όχι μονάχα ορισμένες χώρες μας να είναι μέσα στα πλαίσια αυτής της ομάδας. Διαδικασία catch the eye τώρα. Δεν θα έχουμε χρόνο για όλους γιατί πρέπει να ψηφίσουμε. Θα δώσω το λόγο σε έξι άτομα και μόνο. Ο κύριο Τζίζιπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση για τον Νότιο Κάφκασο είναι μια καλή πράγματι έκθεση. Να υπογραμμίσω και τον ρόλο τον οποίο αναγνωρίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ενδιάμεση και σαν μονάδα που θα προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της περιοχής. Παρ' όλα αυτά κάποια προβλήματα παραμένουν σε κρεμότητα όπως το θέμα της εδαφικής ακαιρεότητας των χωρών αυτών. Θα πρέπει οι χώρες αυτές επίσης να ενισχυθούν οικονομικά και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σταθεί αρρωγός. Υπάρχει το πολύ σημαντικό θέμα επίσης των προσφύγων, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πόσελτ αν δεν μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα των πληθυσμών αυτών, αυτό θα είναι μεγάλη ντροπή για μας. Επίσης θα πρέπει να γίνει αναφορά και στη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Μειονοτήτων. Ευχαριστώ κύριε Γκρτζιπ. Ο κύριος Πάσκο έχει το λόγο. Σήμερα Συζητάμε μία πολύ σημαντική και σωστή έκθεση για μια σημαντική περιοχή. Επίσης αναφέρει γενικά τα της περιοχής η οποία βρίσκεται σε μια στρατηγική τοποθεσία επιτρέπει την ε, μετάβαση αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως έχουν και δικά τους αποθέματα αυτές οι χώρες. Όμως ακριβώς λόγω της στρατηγικής της σημασίας αποτελεί αντικείμενο αντιπαλότητας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και βλέπουμε έτσι τις πολλές παγωμένες ε, συγκρούσεις που επικρατούν ε, εκεί πέρα. Και θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς σε αυτά τα οποία λέμε και κάνουμε έστω και αν δυσαρεστούμε κάποιους και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια στρατηγική. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Βάτσον. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω τον κύριο Κύριλοφ και τον κύριο Καζάκ για το έργο τους. Αν δούμε τις σχέσεις μας μόνο μέσα από το πρίσμα της ανάγκης μας για φυσικό αέριο και πετρέλαιο θα εντείνουμε τις, θα οξύνουμε τις αντιθέσεις και θα αποτύχουμε να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα. Είναι απαραίτητη η ειρήνη και η οικονομική ανάπτυξη στον Νότιο Κάφκασο που πρέπει να είναι η οδηγή της ε, πολιτικής μας θα πρέπει να είναι σε συνεργασία με τις χώρες αυτές στο ΝΑΤΟ για λόγους ασφαλείας. Επίσης θα πρέπει να συνεργαστούμε με τη Ρωσία και την Τουρκία για να μεγιστοποιήσουμε την ισχύ των συμφωνιών και να δώσουμε μια χείρα βοηθείας προς τις χώρες αυτές με διαδικασίες ελευθέρου εμπορίου και προξενικές διευκολύνσεις προξενικών θεωρήσεων. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται και τι έγινε και με τον Γιανούκοβιτ και τον Μετβέντεφ για τη Μολδαβία που δείχνει πόσα πράγματα μπορούν να επιτευχθούν σε θέματα διπλωματίας και νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την προσοχή μας στον τομέα της ε, εταιρική σχέσης προς τα ανατολικά τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αναπτύξει μια πλήρη στρατηγική για τα θέματα της Μαύρης Θάλασσας. Ευχαριστώ κύριε Βουάτσοτ. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Κυρίλοφ και να κάνω κάποια σχόλια για αυτή την έκθεση. Πρώτα απ' όλα η δημοκρατία. Όπως είπε ο κύριος Πόσελ, οι χώρες περιοχής πρέπει να συνεργαστούν. Οι χώρες αυτές μπορούν να συνεργαστούν, το Ζερβαϊτζάν, Γεωργία και η Αρμενία καθώς είναι χώρες όπου ε, υπάρχει κράτος δικαίου. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ωφεληθεί. Το δεύτερο θέμα βέβαια αφορά την ενέργεια. Θα ήθελα να επισημάνω το σημαντικό ρόλο της Γεωργίας και του Αζερβαϊτζάν ως ε, σημείο διέλευσης ε, πηγών ενέργειας και, και Βεβαίω πήγαν ενέργειας και των δύο των χωρών. Οπότε είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια όταν μιλάμε για τη μεταφορά τη ενέργεια από την Αρμενία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο έχει ο κ. Μέλτσερ. Um Κύριε Πρόεδρε, οι ανάγκες να περιορίσουμε την ενεργειακή μας εξάρτηση από την Ρωσία θα πρέπει να είναι οδηγός της πολιτικής μας για τον Νότιο Κάφκασο. Ο Νότιος Κάφκασος παίζει ένα κομβικό ρόλο στην περιοχή αυτή. Δεν είναι μονάχα ένας χώρος διαμετακόμισης για την ενέργεια και το φυσικό αέριο αλλά είναι ένα χώρο ο οποίο είναι κομβικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και για την Τουρκία. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να συνάψουμε συμφωνίε σταθεροποίηση και εταιρική σχέση. Αυτό η σταθεροποίηση στην περιοχή αυτή είναι προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε αυτό το ρόλο όμω μονάχα στην Τουρκία, αλλιώ θα δημιουργήσουμε νέε εξαρτήσει. Όπω έχει φανεί και με το παράδειγμα της Κύπρου, δεν μπορούμε πάντα να βασιζόμαστε σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δώσουμε την ε, υποστήριξή μας στην ε, συμπλήρωση, στην επίτευξη του στόχου της δημιουργίας του αγωγού Ναμπούκου που εδώ για πάρα πολύ καιρό ώστε να μην χαθούν οι πόροι του Νοτιού Καυκάσου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μέλσερ. Κύριος Πάσχας. Κύριε Επίτροπε, Όπως φάνηκε χθε από τους ε, εκπροσώπους της ε, Αρμενίας, τονίσανε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια στρατηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Κάφκασο και θα πρέπει <clears throat> να υπάρξει και στην περίπτωση του Ναγκόνο Καραμπάχ μια κοινή θέση που να συμβαδίζει με αυτά τα οποία ανέφεραν οι χώρες του, του ΟΑΣΕ. Αυτά τα οποία λέγονται όμως στο άρθρο 8 αυτής της, ε, ε, της δήλωσης δεν συμβαδίζουν με αυτά που λέει η δήλωση της Μαδρίτης και η άποψη της ομάδας του Μίνσκ. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να αποτελέσουν ένα εμπόδιο για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στον Αγκόνο Καραμπάχ. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να άρουμε τις επιφυλάξεις μας και στην περίπτωση αυτή να προσπαθήσουμε να βρούμε συμβιβασμούς και να καθυστερήσουμε την ψήφιση αυτής της έκθεσης ώστε οι αρμένοι φίλοι μας να μπορούν να παρουσιάσουν καλύτερα τη θέση τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πάσκα. Ο κύριος Επίτροπος έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιόπτυγμα μέλη. Ο τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Πάσκα, Uh, Είπε κάτι πολύ σημαντικό. Σας παρακαλώ ησυχία. Ο Επίτροπος, θα ήθελα να κάνω κάποιες πολύ σύντομες παρατηρήσεις γιατί ο χρόνος πιέζει. Πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ πως έχουμε στρατηγική και η στρατηγική είναι μέσω της ανατολικής εταιρικής σχέσης οι χώρες αυτές να έρθουν πιο κοντά στην Ένωση και μάλιστα αναφέρεται όσο πιο κοντά γίνεται. Δεύτερον, νομίζω πως έχουμε μέσα για αυτό. Αυτά τα μέσα είναι οι συμφωνίες σύνδεσης, συμφωνίες οικονομικής ε, ολοκλήρωσης, η κινητικότητα, το ζήτημα της βίζας και τέλος μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα συνδυάζει την κοινοτική μέθοδο με την μέθοδο της κοινή πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Και η τρίτη μου παρατήρηση είναι πως αναμένω τις συζητήσεις με τους βουλευτές για το πακέτο γειτονία όπου θα μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα του εάν η έννοια αυτή όσο το δυνατόν πιο κοντά στην Ένωση δηλαδή πρέπει να έχει κάποιον θεσμικό ορισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τον λόγο έχει ο εισηγητής ο κύριος Κύριλοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα σχόλια και για την επικοδομητική συνεργασία. Σας ευχαριστώ για την στήριξη που είχα από την πλειοψηφία των συναδέλφων θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Καζάκ για τις επικοδομητικές ιδέες που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή του και τη συνεισφορά της Επιτροπής Ήτρε, πολλά από τα σημεία της οποίας Βεβαίω, ενσωματώθηκαν στην έκθεση. Ευχαριστώ και την γραμματεία τη Επιτροπή Εξωτερικών για του διάφορου ειδικού και τη ΜΚΟ που συνεισέφεραν επίση και θα ήθελα να πω κάτι. Πρέπει να εφαρμόζουμε τις ίδιες αρχές παντού. Άσκησα άκουσα κάποια κριτική από κάποιους συναδέλφους, πρέπει να ξέρουμε πως ε, κάποιοι λένε πως δεν θα μας υποστηρίξουν εάν μιλήσουμε για αυτοδιάθεση και εδαφική αικαιρεότητα της γεωργίας θεωρούν πως αυτή είναι η καλύτερη ε, αρχή για να οικοδομήσουμε τις σχέσεις μας. Ελπίζω το Συμβούλιο και η Κομισιόν να ακούσουν τις συστάσεις του Κοινοβουλίου και να καταλήξουν σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική της Ένωσης για τον Νότιο Κάφκασο και βεβαίως θα ήθελα να επισημάνω πως ο κύριος Φούλε, ο Επιτροπός, επισκέφθηκε σε πολύ κρίσιμη στιγμή την Επιτροπή. Επίσης να απευθύνω έκκληση στην Βαρόνια Άστον να κάνει το ίδιο και να προσπαθήσει να προλάβει τις συγκρούσεις στην περιοχή καλωσορίζουμε και στηρίζουμε την απόφαση της προηγούμενης εβδομάδας του Συμβουλίου να υιοθετήσει οδηγίες ε, για τις συμφωνίες σύνδεση με τις τρεις χώρες και θεωρούμε πως η αναβάθμιση των σημαντικών σχέσεων με τις τρεις χώρες είναι σημαντικό βήμα. Έχει φτάσει η στιγμή να προσπαθήσουμε περισσότερο να μην κλιμακωθούν οι εντάσεις και τα προβλήματα στην περιοχή, αλλιώς κινδυνεύουμε να παρεμβούμε πάλι και δεν θα πρέπει να περιμένουμε να είναι πάρα πολύ αργά. Το μεγάλο μάθημα που έμαθε η Ευρώπη είναι το μάθημα της ολοκλήρωσης. Είναι ο μόνος βιώσιμος τρόπος συμφιλίωσης με το παρελθόν και επένδυση στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο Πρόεδρος θα κάνει μια ανακοίνωση και θα συνεχίσουμε με την ψηφοφορία αμέσως μετά.